ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Now we hear the... Κύριε Πρόεδρε της Τσεχικής Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να σε απευθύνω θερμότατο χαιρετισμό. Σας εύχομαι το καλό ορίσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των εκπροσώπων των, ε, των εκλεγμένων εκπροσώπων των ευρωπαϊκών λαών. Η χώρα σας, κύριε Πρόεδρε, πάντοτε βρέθηκε στην καρδιά της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ήδη από τον 14ο αιώνα ο Κάρολος ο καρολος ο ως αυτοκράτορ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έκανε την Πράγα πρωτεύουσά του. Θυμούμεθα ότι ο βοημός βασιλέας Γιώργιος ήταν μεταξύ των πρώτων μεγάλων Ευρωπαίων και ήδη από το 1462 καταβάλει προσπάθειες για την δημιουργία μιας ένωσης κρατών. Συνεχίζοντας την παράδοση της χώρας σας, εκτιμούμε και σήμερα τον σημαντικό ρόλο της τσεχικής δημοκρατίας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η τσεχική δημοκρατία που παίζει σημαντικό και ενεργό ρόλο ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήδη. Από τις πρώτες μέρες της η τσεχική προεδρία κρίθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Τον πόλεμο στη Γάζα, την κρίση του φυσικού αερίου που οδήγησε ώστε 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στερηθούν την προμήθεια ενέργειας. Η Τσεχική Προεδρία και ιδίω ο Πρωθυπουργός σας, Μιρέκ Τοπολάνεκ, καθώς και ο Υπουργός σας των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αναπληρωτής Πρωθυπουργός, Αλέξανδρος Βοντράν, ο οποίος είναι εδώ παρόν και το απευθύνω επίση χαιρετισμό, όπως επίσης και ο Υπουργός των Εξωτερικών, Κάρολ Σβάλτσενμπεργκ, έχουν παίξει θετικότατο ρόλο. Σήμερα η τσεχική δημοκρατία φέρει μεγάλη ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω την τσεχική δημοκρατία και να την συγχαρώ, διότι την Τετάρτη το τσεχικό κοινοβούλιο εκύρωσε με μεγάλη πλειοψηφία την συνθήκη της Λισαβόνας. η ψηφοφορία αυτή υπογραμμίζει την διάθεση της Προεδρίας για θετική πρόωθηση της περαιτέρω διαδικασίας κυρώσεως και για την συμβολή στην επιτυχία της νέας συνθήκης που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άκουσε και σημείωσε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις προγραμματικές δηλώσεις της Τσεχικής Προεδρίας. Και η συνδιάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων που οργανώθηκε τούτην εδώ την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συμμετοχή του βεβαίως, με το θέμα ένα New Deal για την ευρωπαϊκή ανοικοδόμηση της οικονομίας δηλαδή έχει μεγάλη σημασία. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι σαφείς εθνικές προστατευτικές τάσεις είναι ανισχυτικές. Οφείλουμε να αντισταθούμε και να αντιταχθούμε σε αυτές, διότι όλοι έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε την ενιαία αγορά από την οποία όλοι υποφελούμεθα. Οι ελπίδες μας επαφιένται σε εσά, στην τσεχική δημοκρατία και σε εσά κύριε Πρόεδρε, που είστε γνωστός ως υποστηρικτής και οπαδός μιας ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Ένα παλιό γνωμικό της ε, Βοημίας λέει ότι είναι καλύτερα να διαπραγματεύεται κανείς επί μια διετία παρά να κάνει πόλεμο για δύο εβδομάδες. Όλοι κατανοούμε βεβαίως εσάς κύριε Πρόεδρε καθώς και τους πολίτες της χώρας σας που τάσσονται υπέρ της συμφιλίωσης και της διαβούλευσης και που εμείς έχουμε κάνει πραγματικότητα τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Εν προκειμένου και οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου έχουν μέγιστη σημασία. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε όπου όπως είπατε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά σας προς τους Τσέχους πολίτες τους καλέσατε να προσέλθουν πολυάριθμοι και να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εύχομαι στην Τσεχική Δημοκρατία επιτυχή και καρποφόρο Τσεχική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα να μιλήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ένα από τα, από τα όργανα κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω έρθει κάμποσε φορέ εδώ, ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω στην Ολομέλεια. Γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόσκλησή σας. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι 27 χωρών με σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων είναι ένα μοναδικό ακροατήριο. Τόσο μοναδικό και στην ουσία του και τόσο επαναστατικό όσο το ίδιο το πείραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πάνω από 50 χρόνια η Ένωση προσπάθησε να βελτιώσει το σύστημα λήψεων αποφάσεων στην Ευρώπη μετακινώντας ένα σημαντικό τμήμα των αποφάσεων από τα κράτη-μέλη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έρχομαι εδώ από την πρωτεύουσα της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας, την Πράγα, από το ιστορικό κέντρο της ε, Τσεχοσύνης, από ένα από τα σημαντικά μέρη όπου Βόηθησε να αναδυθεί η ευρωπαϊκή σκέψη, η ευρωπαϊκή κουλτούρα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Έρχομαι ως εκπρόσωπος του τσεχικού κράτους, που ανέκαθεν και με διάφορες μορφές υπήρξε τμήμα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Έρχομαι από ένα κράτος το οποίο πολλές φορές πήρε άμεσο και σημαντικό μέρος στη διαμόρφωση της ιστορίας και θέλει να εξακολουθήσει να το κάνει. Πριν από εννέα χρόνια ήταν πριν από εννέα χρόνια που τελευταία φορά ο πρόεδρος τη Τσεχική Δημοκρατία σα μίλησε. Πρόκειται για τον προκάτοχό μου, Βάτσλακ Χάβελ. Και αυτό τέσσερα χρόνια πριν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν μερικές εβδομάδες, ο πρωθυπουργό της Τσεχίας, Μίρεκ Τοπολάνεκ, επίσης, και αυτό σας μίλησε, ως ηγέτης μιας χώρας που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ένωσης η ομιλία του εστιάστηκε στις προτεραιότητες της ψυχικής Προεδρίας όπως επίσης και σε επίκαιρα προβλήματα που, αντιμετωπίζει σήμερα, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι, ευρωπαϊκές, οι χώρες της Ένωσης. Αυτό μου επιτρέπει με τη σειρά μου να επικεντρωθώ σε θέματα που είναι κάπως πιο γενικά. Θα ήθελα να σας μιλήσω για θέματα που από μια πρώτη ματιά ίσως φαίνονται λιγότερο σημαντικά όσο το να επιλύσουμε την τρέχουσα οικονομική κρίση ή το, η αντιπαράθεση όσον αφορά το αέριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ή η κατάσταση στη Γάζα. Ωστόσο, θεωρώ ότι και αυτά τα θέματα είναι άκρα σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης λιγότερους από τρεις μήνες η Τσεχική Δημοκρατία θα εορτάσει την επέτειο της πέμπτης, του πέμπτου έτους από την ένταξή της στην Ένωση. Αυτό θα το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Αυτό θα το γιορτάσουμε σαν μια χώρα η οποία σε αντίθεση με ορισμένες άλλες νέες χώρες μέλη δεν αισθάνεται απογοητευμένη από, λόγω ανεκπλήρωτων προσδοκιών που συνδεόταν με τη συμμετοχή μας στην Ένωση. Αυτό δεν πρέπει να εκπλήσει, διότι υπάρχει μια λογική εξήγηση γι' αυτό. Οι προσδοκίες μας ήταν ρεαλιστικές. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα μπαίναμε σε μια κοινότητα που διαμορφώνεται από ανθρώπους. Ξέραμε ότι δεν ήταν ένα ουτοπιστικό οικοδόμημα, Πρόκειται για ανθρώπινο συμφέροντα, ανθρώπινα οράματα, απόψεις και ιδέες. Όλα αυτά τα συμφέροντα και οι ιδέες ε, βρίσκονται σε όλη την Ένωση. Και αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εμείς θεωρήσαμε την ένταξή μας στην Ένωση αφενός ως μια επιβεβαίωση του γεγονότος ότι σχετικά γρήγορα, σε λιγότερα από 15 χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού, καταφέραμε και πάλι να γίνουμε μία μέση ευρωπαϊκή χώρα παρόμοια με τις άλλες. Απ' την άλλη, θεωρήσαμε αυτό σαν μια ευκαιρία να πάρουμε μέρος στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης, σαν μια ευκαιρία να υποφεληθούμε από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήταν ήδη αρκετά προωθημένο και ταυτόχρονα να επηρεάσουμε τη διαδικασία αυτή με βάση τις απόψεις μας αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας όσον αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτό το αίσθημα ευθύνης προσεγγίζουμε και το θέμα της προεδρίας μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι οι πρώτες έξι εβδομάδες της Τσεχικής Προεδρίας πιστικά απέδειξαν την υπεύθυνη αυτή στάση μας. Από αυτό το βήμα επαναλαμβάνω τη βαθιά μου πεποίθηση και το λέω ανοιχτά και με σαφήνεια για όσους από εσά δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να ξέρετε. Η πεποίθησή μου είναι ότι για μας ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει σημαντική πολιτική δύναμη στη χώρα μου που θα ήθελε ή θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτή τη θέση. Συνεπώς, μας συγκινεί ιδιαίτερα το θέμα των συχνών επαναλαμβανόμενων και αυξανόμενων επιθέσεων κατά της χώρας μου που στηρίζεται στην αβάσιμη υπόθεση ότι οι Τσέχοι προσπαθούν να βρουν ένα άλλο είδος σχέδιο ενσωμάτωσης και όχι αυτό που είχαμε κατά νου όταν γίναμε μέλη πριν από πέντε χρόνια. Αυτό δεν αληθεύει. Οι πολίτες της τσεχικής δημοκρατίας θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει μια σημαντική αποστολή που θα μπορούσα να την συνοψίσω ως εξής. Πρώτο, να αρθούν εμπόδια μη αναγκαία και αρνητικά για την ελεύθερη ελευθερία, την ευημερία, την ελεύθερη κυκλοφορία των λαών, των προϊόντων, των υπηρεσιών, των ιδιών, των πολιτικών φιλοσοφιών, των κοσμοθεωριών, των πολιτιστικών μορφών και διαφόρων μοντέλων συμπεριφοράς που επικρατούν στην Ευρώπη εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερον, μια κοινή φροντίδα για τα δημόσια αγαθά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρουμε σε προγράμματα που δεν είναι δυνατόν αποτελεσματικά να ελοποιηθούν με διμερείς διαπραγματεύσεις δύο ή τριών ας πούμε γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών. Οι προσπάθειες να υλοποιηθούν αυτοί οι δύο στόχοι, δηλαδή να αρθούν τα εμπόδια φενός και λογικά να επιλεγούν θέματα που είναι δυνατόν να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά δεν έχουν συμπληρωθεί και δεν θα συμπληρωθούν ποτέ. Παραμένουν ακόμα εμπόδια και η λήψη των αποφάσεων στο επίπεδο των Βρυξελών σίγουρα είναι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Σίγουρα είναι παραπάνω από ό,τι οι λαοί σε επιμέρους κράτη-μέλη ζητούν. Εσείς, οι Ευρωβουλευτές, σίγουρα το ξέρετε αυτό. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω συνεπώς είναι θεωρητικό. Πιστεύετε πραγματικά ότι κάθε φορά που ψηφίζετε αποφασίζετε κάτι που πρέπει να αποφασιστεί εδώ και όχι πιο κοντά στους πολίτες, δηλαδή στα επιμέρους ευρωπαϊκά κράτη. Με βάση την πολιτικά ορθή φρασιολογία που ακούμε συχνά αυτές τις μέρες, ακούμε και για άλλες ενδεχόμενες επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης που είναι δευτερεύουσα σημασίας. Αυτά κινούνται από τις φιλοδοξίες των επαγγελματιών πολιτιών και ατόμων που συνδέονται με αυτούς και όχι από τα συμφέροντα του μέσου πολίτη των κρατών μελών μας. Όταν είπα ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ούτε δεν έχει μπροστά της άλλη εναλλακτική λύση και το ξανατονίζω αυτό είπα μόνο τα μισά από όσα θα έπρεπε να υποθούν τα άλλα μισά λογικά της δήλωσής μου είναι τα εξής οι μέθοδοι και οι μορφές ευρωπαϊκής ενοποίησης αντίθετα έχουν πάρα πολλές διαφορετικές θεμητές μορφές, εναλλακτικές μορφές. Η ιστορία δεν σταματάει ποτέ, όπως είδαμε το τελευταίο μισό αιώνα. Το να πούμε ότι το status quo, δηλαδή η σημερινή θεσμική μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα δόγμα πέραν πάσης κριτικής, υπεράνω κριτικής, είναι λάθος, που δυστυχώς παρόλα αυτά διαδίδεται και κυκλοφορεί. Αν και έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση όχι μόνο με τη λογική σκέψη αλλά και με την δυσχυλιετή ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το ίδιο λάθος συμβαίνει και με υποθέσεις απριόρι χωρίς να έχει υποστεί κριτική υπόθεση ότι υπάρχει μόνο ένα δυνατό και σωστό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση που είναι η Ένωση να είναι όλο και πιο συνεκτική Ever Closing Union δηλαδή μια πρόοδος προς όλο και βαθύτερη πολιτική ενοποίηση των κρατών μελών αλλά ούτε το σημερινό status quo ούτε η υπόθεση της συνεχούς εμβάθυνσης της ενοποίησης είναι κάτι το θετικό και θα δεν θα έπρεπε να είναι δόγμα για κανέναν Ευρωπαίο Δημοκράτη. Όλες αυτές οι έννοιες προωθούνται από ορισμένους που αυτοανακηρύσσονται, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του φημισμένου συγγραφέα από τη Τσεχία Μίλα Κούντερα. Αυτοανακηρύσσονται λοιπόν οι κλειδοκράτορες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μία τέτοια προσπάθεια είναι απαράδεκτη. Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι οι διάφορες θεσμικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι ένα εργαλείο για την υλοποίηση των ουσιαστικών στόχων. Η ουσιαστική αυτή στόχη είναι η ανθρώπινη ελευθερία και ένα οικονομικό σύστημα που θα εξασφαλίζει την ευημερία. Και το σύστημα αυτό είναι η οικονομία της αγοράς. Είμαι βέβαιος ότι αυτό προσδοκούν οι πολίτες όλων των χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, τα 20 χρόνια που ακολούθησαν την κατάρρευση του κομμουνισμού, έχω γίνει επανειλημμένος μάρτυρας του γεγονότος ότι τα αισθήματα και οι φόβοι είναι περισσότεροι από αυτός που πέρασαν ένα τμήμα του 20ου αιώνα χωρίς την ελευθερία και έδωσαν μάχη υπό ένα κεντροσχεδιασμένο δυσλειτουργικό καθεστώς. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι ε, σε οποιοδήποτε φαινόμενο και τάση που οδηγεί σε άλλη κατεύθυνση από αυτή της ελευθερίας και της ευημερία. Και οι πολίτες της τσεχικής ε, δημοκρατίας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το παρόν σύστημα λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικό από ένα, από ένα σύστημα κλασικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως έχει δοκιμαστεί στην ιστορία. Σε ένα κανονικό κοινοβουλευτικό σύστημα, ένα τμήμα των βουλευτών υποστηρίζουν την κυβέρνηση και ένα άλλο τμήμα την αντιπολίτευση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει τέτοια διευθέτηση. Εδώ υπάρχει μόνο μία εναλλακτική λύση που προωθείται. Και όσοι τολμούν να τάσσονται υπέρ μια άλλη τάση, σημαδεύονται ως εχθροί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σχετικά πρόσφατα, στο δικό μας τμήμα της Ευρώπης, Ζούσαμε κάτω από ένα πολιτικό σύστημα που δεν επέτρεπε εναλλακτικέ λύσεις. Και ω εκ τούτου δεν ανεχόταν την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Μέσω αυτής της εμπειρίας διδαχθήκαμε το πικρό μάθημα ότι χωρίς αντίθεση, χωρίς αντιπολίτευση δεν υπάρχει ελευθερία. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές ε, εναλλακτικές λύσεις. Και όχι μόνο αυτό. Η σχέση μεταξύ του πολίτη ενός κράτους και του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μια συνηθισμένη σχέση όπως μεταξύ ενός ε, ψηφοφόρου και ενός ε, πολιτικού που τον εκπροσωπεί. Μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια τεράστια απόσταση και όχι μόνο από γεωγραφική άποψη. Η απόσταση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντίστοιχη στις χώρες μέλη και αυτή η απόσταση έχει χαρακτηριστεί πολύ συχνά ως δημοκρατικό έλλειμμα, έλλειψη δημοκρατικής λογοδοσίας και λήψη αποφάσεων όχι από τους εκλεγμένους, από τους επιλεγμένους, η υπερβολική γραφειοκρατικοποίηση. Οι προτάσεις ε, για τη μεταρρύθμιση του Στάτου Κβό που συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που έχει απορριφθεί ή στην παρόμοια συνθήκη της Λισαβόνας θα επιδίνωναν αυτό το ελάττωμα το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Έθνος, το ελάττωμα αυτό, το έλλειμμα αυτό, δεν μπορεί να επιληθεί μόνο από την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αντίθετα θα επιδεινώσει το πρόβλημα και θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αποξένωση, αλλοτρίωση μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Η λύση δεν θα ήταν να προσθέσουμε λάδι, καύσιμο στο καζάνι αυτού του τύπου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή να καταργήσουμε το ρόλο των κρατών μελών στο βοβό μιας νέας ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών που θα είναι πολυεθνική και πολυπολιτισμική. Τέτοιου τους απόπειρε έχουν ε, αποτύχει συστηματικά στο παρελθόν γιατί δεν αντανακλούσαν τις αυθόρμητες ιστορικές εξελίξεις. Πολύ φοβούμε ότι οι απόπειρες αυτές να επιταχυνθεί και να εμβαθυνθεί η ολοκλήρωση και να μετατεθούν οι αποφάσεις για τις ε, ζωές των πολιτών από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τέτοιες απόπειρες θα έχουν επιπτώσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο όλα τα θετικά επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, την τελευταία πεντηκονταετία. Ας μην υποτιμούμε τους φόβους των πολιτών πολλών χωρών μελών που ανησυχούν ή φοβούνται ότι τα προβλήματά τους τα αποφασίζουν ερήμην τους, άλλοι μακριά από αυτούς και η δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να επηρεάσουν αυτές τις αποφάσεις είναι πολύ περιορισμένη. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επιτυχής εν μέρη χάρη στο γεγονός ότι η ψήφος κάθε χώρας έχει το ίδιο βάρος με τις υπόλοιπες και άρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί να αγνοηθεί. Να μην επιτρέψουμε να διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου οι πολίτες των χωρών μελών θα ζουν τη ζωή τους ε, με την αίσθηση ότι το ευρωπαϊκό όραμα δεν είναι δικό του όραμα και ότι έχει πάρει στραβή κατεύθυνση, τελείω διαφορετική από αυτή που προσδοκούσαν και απλώ του επιβάλλεται ερήμην του. Γιατί πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα θα ολιστήσουμε προς εποχές που ελπίζαμε ότι θα ανήκαν πια στην ιστορία. Το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το θέμα της ευημερία. Θα πρέπει να πούμε απερίφραστα ότι το παρόν οικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σύστημα καταπιεσμένης αγοράς με μόνιμες προσπάθειες ενίσχυσης της, κεντρο... της κεντροελεχόμενης οικονομίας. Και παρόλο που η ιστορία μας έχει αποδείξει καθαρά και ξεάστερα ότι μια τέτοια μέθοδος οδηγεί σε διέξοδο, παρόλα αυτά φαίνεται ότι ακολουθούμε το ίδιο μονοπάτι. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια κυβερνητική προσπάθεια μόνιμης περικοπής της αυθόρμητης ε, διαδικασίας της αγοράς. Και τους τελευταίους μήνες είχαμε ταυτόχρονα πολύ εσφαλμένη ερμηνεία για τα αίτια της παρούσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης θεωρούμε υπέτειο την ελεύθερη αγορά για την κρίση αυτή, ενώ στην ουσία πρόκειται για ακριβώς το αντίθετο. Η πολιτική χειραγώγηση της αγοράς οδήγησε στην χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει και πάλι να θυμηθούμε την ιστορική εμπειρία της δικής μας ε, ευρωπαϊκής περιοχής και να θυμηθούμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Πολλοί από εσά θα γνωρίζετε το όνομα του Γάλλου οικονομολόγου Φρεντερίκ Μπαστιά, ενός οικονομολόγου του 19ου αιώνα και τη γνωστή του Petition of the Candlemakers που έχει γίνει ένα κλασικό ανάγνωσμα της οικονομίας και απέδειξε την ουτοπία της πολιτικής επέμβασης στην οικονομία. Στις 14 Νοεμβρίου του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μία πραγματική και όχι μία εικονική τέτοια πρόταση και επέβαλε ένα, δεσμό ε, δασμό 66% στα εισαγόμενα από την Κίνα κεριά. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι ένα έγγραφο 160 χρόνων θα γινόταν επίκαιρο και θα εφαρμοζόταν τη σήμερα ημέρα. Και όμως συνέβη αυτό. Ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της εκτετικής εφαρμογής τέτοιων μέτρων στην Ευρώπη είναι μια οικονομική επιβράδυνση, για να μην πω μια πλήρης αναχέτηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η μοναδική λύση είναι η απελευθέρωση και η απορρίθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς, της ευρωπαϊκής οικονομία Και σας τα λέω όλα αυτά γιατί αισθάνομαι μια τεράστια ευθύνη για την εξασφάλιση της ε, δημοκρατικής και ευήμερης Ευρώπης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις στοιχειώδεις αρχές που για αιώνες αποτέλεσαν τους ε, ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού πολιτισμού, για να μην πω για χιλιετίες. Είναι αρχές που έχουν διαχρονική αξία, είναι οικουμενικού χαρακτήρα και θα πρέπει να ακολουθηθούν και από την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πολίτες των χωρών μελών επιθυμούν ελευθερία, δημοκρατία και οικονομική ευημερία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το πιο σημαντικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ελεύθερη συζήτηση για όλα αυτά τα προβλήματα. Να μην φημωθεί μια τέτοια ελεύθερη συζήτηση ως επίθεση της ίδιας της ουσίας ε, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είμαστε ανέκαθε της γνώμη ότι η ελεύθερη συζήτηση για τόσο σοβαρά θέματα, η δυνατότητα έκφρασης της γνώμης, η προάσπιση του δικαιώματος ε, οποιοδήποτε να εκφράσει μια άποψη που διαφέρει από την κρατούσα άποψη, άσχετα και διαφωνούμε με αυτή, είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και μια τέτοια αρχή την είχαμε στερηθεί για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Εμείς που περάσαμε ακούσει από μια τέτοια εμπειρία που μας δίδαξε ότι μια ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών είναι η βασική προϋπόθεση μιας υγιούς δημοκρατίας εμείς λοιπόν ελπίζουμε ότι η προϋπόθεση αυτή θα τηρηθεί και θα γίνει σεβαστή και στο μέλλον. Αυτή είναι η ευκαιρία και η μοναδική μέθοδος για να δημιουργήσουμε μια πιο ελεύθερη, πιο δημοκρατική και πιο ευήμερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Πέτερινγκ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε της Τσεχικής Δημοκρατίας, επιθυμία σας ήταν να μπορέσετε να λάβετε το λόγο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαρίστως δεχτήκαμε να εκπλώσουμε την επιθυμία σας. Σε ένα κοινοβούλιο του παρελθόντος, ασφαλώς δεν θα μπορούσατε να είχατε εκφωνήσει παρόμοιο λόγο. Δόξα τω Θεώ, ζούμε σήμερα σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία όπου καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε μια ευρωπαϊκή οικογένεια και όπως σε κάθε οικογένεια υπάρχουν και διαφορές απόψεων. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε και μόνο λίγα σχόλια θα κάνω, αλλά νομίζω ότι έχω και την υποχρέωση να το πράξω. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων. Μια κοινότητα ανθρώπων χαρακτηρίζεται από το ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα, ισχυρά σημεία, αδυναμίες και οφείλουμε να κάνουμε κοινή προσπάθεια για να ενισχύσουμε τα δυνατά μας σημεία και να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες μας. Και συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν κάθε απόφαση που λαμβάνουμε θα μπορούσε να έχει ληφθεί αλλού. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το θέσουν το ερώτημα και οι πρωτεύουσε των κρατών μα. Μήπω ορισμένε αποφάσει πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα στο τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και όχι στο επίπεδο των πρωτεύουσών των κρατών. Και επιτρέψτε μου μια τελική παρατήρηση η οποία έχει σχέση και με την αυτοσυνείδηση του Κοινοβουλίου μας. Σας ευχαριστούμε για την αναγνώριση, για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντικό θεσμό. Εάν σήμερα δεν διέθετε την επιρροή που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν δεν ήμασταν σήμερα συνομοθέτης στο 75% των περιπτώσεων και εάν κυρωθεί εν τέλει η συνθήκη της Λισαβόνας θα είμαστε σχεδόν για το 100% συνομοθέτες. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, θα αποφάσιζε η γραφειοκρατία στην Ευρώπη, αλλά τώρα αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας που αποτέλεσε έκφραση της ποικιλία απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και στην Δημοκρατία εν τέλει ισχύει η άποψη της πλειοψηφίας. Και τασόμαστε υπέρ της ελευθερίας, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ τούτης εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.